Ε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ε, σας παρακαλώ να συγχωρέσετε την καθυστέρηση, αλλά ο συνήθως, αυτό είναι αναπόφευκτο, κάθε χρόνο, γιατί για να προετοιμάσουμε αυτή τη ψηφορία που είναι δύσκολη και χρονοβόρα ε, για τις τροπολογίες του προπολογισμού του προσεχούς έτους Έχω, υπάρχει ανάγκη να οριστικοποιήσουμε μια πολιτική συμφωνία όσο το δυνατόν πληθρέστερη μεταξύ όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτικών ομάδων. Ε, γι' αυτό ο εισηγητής ε, δούλεψε μαζί με τους σκιώδεις της κάθε ομάδας και τη γραμματεία την οποία θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω για την πραγματικά θαυμάσια εργασία που έκαναν και σήμερα το πρωί χρειαστήκαμε δύο ολόκληρες ώρες για να δούμε τις λεπτομέρειες των σημείων συμφωνίας και να διευκρονίσουμε τα σημεία που δεν επιτεύχθηκε συμφωνία. Ε, Χαιρετώ την παρουσία του Γενικού Διευθυντού της Επιτροπής. Τον ευχαριστώ και θα έχει ασφαλώς την ευκαιρία να πάρει το λόγο. Πρώτο σημείο, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν ε, παρεμβάσεις, θεωρείται ε, ότι εγκρίνεται. Δεύτερο σημείο, η έγκριση των πρακτικών της συνάντησης της 22ης Σεπτεμβρίου. Εγκρίνεται λοιπόν εγκρίνονται και τα πρακτικά. Στα Κοκομπού θα είδατε τις ε, πληροφορίες ε, που έδωσε ο Πρόεδρος ε, στο σημείο 3. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να επανέλθω. Θα ήθελα να προσθέσω μια άλλη πληροφορία στη συνάντηση των συντονιστών της περασμένης εβδομάδας αποφασίστηκε η συνέχεια της απόφασης διάσκεψης των Προέδρων σε σχέση με τη σύνθεση των αντιπροσωπιών του Κοινοβουλίου που θα διαπραγματευτεί μαζί με την ε, Τρόικα της ε, Προεδρίας του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε η αντιπροσωπή αυτή να συσταθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στον Προϋπολογισμό, επικεφαλής της και τους δύο συνεισηγητές για τις δαπάνες και για τους δύο εισηγητές για τα έσοδα. Άρα λοιπόν η συνάντηση των συντονιστών της ε, περισμένης εβδομάδας αποφάσισε όμως ότι για τις δαπάνες θα είναι ο Ράιμαρ Μπέργκε, ο οποίος ε, θα έχει τον τίτλο του Γενικού Εισηγητού και θα υπάρξει ένας δεύτερος εισηγητής που είναι ο συνάδελφός μας Ήβαλο Καλφίν, ο οποίος ε, δεν μπορεί να σήμερα γιατί έχει έντονες πολιτικές δραστηριότητες στη χώρα του και ανάλογα με τις ε, πολιτικές εξελίξεις εμείς ε, ελπίζουμε από εγωιστική άποψη, εγωιστικά καθαρά να παραμείνει συγκητής. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τα έσοδα, ο Ζαν Λουίκ Ντεάν με την ε, συνδρομή του Άνιεσεν συγκητή. Euh, την κυρία Άνισεν, λοιπόν, που θα ασχοληθούν με το θέμα της ε, χρηματοδότησης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης σε σχέση με κάποιες ε, μειώσεις. Τώρα, όσον αφορά, και έρχομαι στο σημείο 4, όσον αφορά την οργάνωση της ψηφοφορίας, έχουμε θέσει ένα στόχο ο οποίος νομίζω ότι θα ικανοποιήσει όλα τα μέλη και που είναι να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία αύριο το βράδυ στις, στις 6.30. Συγγνώμη. Έχουμε προβλέψει ως πολιτικό μέτρο, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο, τη δυνατότητα βεβαίως να έχουμε ένα επιπλέον πρωί της Πέμπτης αν χρειαστεί. Έχουμε την εντύπωση ότι ο πολιτικός διάλογος έχει αρκετά προχωρήσει μεταξύ των πολιτικών ομάδων, ώστε να μπορούμε να πάμε αρκετά γρήγορα με την ψηφοφορία, να κρυθούμε γρήγορα. Άρα λοιπόν ο στόχος μας, ο στόχος που έχουμε ορίσει, που ορίσαμε σήμερα το πρωί στη συνάντηση των ε, συντονιστών, είναι να αφιερώσουμε το τέλος του πρωινού σε μια εξέταση της κατάστασης των, της πολιτικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των πολιτικών ομάδων ε, στη βάση των παρουσιάσεων των εισηγητών και να ακούσουμε επίσης και το Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με την ε, παράδοση θα εμφανιστεί εδώ και με την ε, σύμφωνη γνώμη των εισηγητών θα πρότεινα να του δώσουμε πρώτα το λόγο ούτε ώστε οι εισηγητές να μπορούν στις παρεμβάσεις του να απαντήσουν ενδεχομένω σε κάποιες ε, απαντήσεις ή παρατηρήσεις του κλπ. Να τοποθετηθούν, εν πάση περιπτώσει. Στη συνέχεια θα έχουμε την πάυση του μεσημεριανού φαγητού για τις ε, διμερείς επαφές μεταξύ εισηγητών και σκιονδών και θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία στις 3 ε, το απόγευμα. Η βασική ιδέα είναι ε, σήμερα το απόγευμα να ψηφίσουμε τις κατηγορίες που φαινομενικά ε, τουλάχιστον γύρουν τα λιγότερο προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι υπάρχει πολιτική συμφωνία αλλά η κάθε πολιτική ομάδα γνωρίζει τι θα ψηφίσει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τουλάχιστον την οργάνωση ψηφοφορία. Και θα δούμε τα αποτελέσματα. Κατηγορίε 1 και 2, α και β, κατηγορία 2 και κατηγορία 3α. Ε, σήμερα το απόγευμα θα ψηφιστούν. Στην ε, αρχή του απογεύματος θα δούμε και σε σχέση με τις με τις ημερείς επαφές ε, κατά τη μεσημβρινή πάυση εάν έχουμε ανάγκη μια νέα συνάντηση των συντονιστών στις 6.30 εάν χρειάζεται να νοσικοποιήσουμε τις πολιτικές συμφωνίες. Και αύριο το πρωί στις 9 θα ψηφίσουμε το πρωί το υπόλοιπο της κατηγορίας 3β, 3, 3β όλη την κατηγορία 4 μαζί με τους αριθμούς και τα σχόλια τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ιδιαίτερα για την κατηγορία 4 και την κατηγορία 5 που αφορά για τον προπολογισμό της Επιτροπής, της δαπάνες λειτουργίας του κυρίου Ζανζουάν τον οποίων θέλουμε κάπως να θέσουμε υποπίεση. Και αύριο το απόγευμα θα έχουμε τη ψηφοφορία για τις ε, κατηγορίες που έχουν μια προτεραιότητα για τις περισσότερες πολιτικές ομάδες, τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις και στη συνέχεια τον προπολογισμό των άλλων θεσμικών οργάνων, την κατηγορία 5 που αφορά τα άλλα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανόμενο και το προπολογισμό του Κοινοβουλίου, γνωρίζοντας ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα ψηφίσουμε παρά μόνο τις γραμμές του προπολογισμού με τους αριθμούς και τα σχόλια και όσον αφορά τα σχέδια ψηφίσματος, η ψηφοφορία θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στις 13 ε, και η προθεσμία για την κατάθεση ψηφοφοριών είναι η 5η 6 του μηνός 6 ε, ώρα. Οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν στα αγγλικά. Ωραία λοιπόν και θα ήθελα να προσθέσω ότι αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε επίσης το σχέδιο έκθεσης του Ιβαλο Καλφίν για τις εγγύησεις και τις ενδεχόμενες ε, απώλειες της Τράπεζας Επενδύσεων για δάνεια που έχουν χορηγηθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θυμάστε αυτή την ιδιαίτερως ε, μακρά διαπραγμάτευση ε, τριμερείς διαλόγους που έγιναν με το Συμβούλιο και τον κύριο Καλφίν και που κατέληξε σε μια συμφωνία η οποία οποία θα υποβληθεί σε ψηφοφορία αύριο το πρωί στις 9. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με αυτήν την ψηφοφορία. Άρα λοιπόν προτείνω στον κύριο Γενικό Διευθυντή να μας κάνει τις δικές του εισαγωγικές ε, δηλώσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να παρέμβω για να παρουσιάσω κάποια σχόλια πριν να περάσετε στην ε, ψηφοφορία για τις τροπολογίες. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι πολλές από αυτές τις τροπολογίες μας βρίσκουν σύμφωνους ε, στο βαθμό που αποκαθιστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό το επίπεδο των ε, πιστώσεων υποχρεώσεων που, που είχε αρχικά ε, προτείνει η Κομισιόν και το Συμβούλιο περιέκοψε στην πρώτη του ανάγνωση. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τις πίστες πληρωμών. Η περικοπή στην οποία προέβη το Συμβούλιο είναι της τάξης του 3,7 δις ευρώ. Είναι σαφές πως είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο γιατί υποθηκεύει σε υπερβολικό βαθμό και αυτό για δεύτερη διαδοχική χρονιά γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τι συνέβη πέρυσι, τον ε, τίτλο, την κατηγορία 1α, δηλαδή τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα, την ε, ανάπτυξη. Όλα δηλαδή όσα θέλουμε να κάνουμε μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 και το εν κατηγορία 1β όπου έχουμε τη συνοχή και την εκτέλεση των διευθυντικών ταμείων πράγμα που είναι κεφαλαιόδης σημασία σε αυτήν την φάση δυσκολίας. Επίσης ε, προχωράμε στην ανάλυση της εκτέλεσης για το 2011 θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε, αλλά θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι αυτή η εκτέλεση θα μπορούσε να είναι πιο ψηλή, πολύ πιο ψηλή από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και κατά συνέπεια Αντίθετα με τα άλλα χρόνια, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πως ε, γενική, το γενικό έμβασμα να μην ανταποκριθεί στις ανάγκες ε, πιστώσεων, πληρωμών που έχουν εντοπιστεί. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε ε, στην ε, συνδιαλλαγή με τα νέα στοιχεία για την εκτέλεση και η συζήτηση θα πρέπει να γίνει από αυτής της βάσης. Αλλά ήθελα να το υπογραμμίσω ήδη εξ αρχής για να το έχετε υπόψη Ανάμεσα στα σε ε, Τροπολογίε που τονίζουν τις προτεραιότητε του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν δύο που θα ήθελα να υπογραμμίσω περισσότερο γιατί πρόκειται για ανησυχίε ε, οι οποίε είναι κοινέ και για την Κομισιόν. Η πρώτη τροπολογία είναι αυτή που σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ε, Διανομή Επισητιστικής βοήθεια για την εξασφάλιση τη δωρεάν, διατροφής, δωρεάν διανομής τροφίμων σε ευρωπαίου πολίτε. Ξέρετε πόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον τελευταίο καιρό για ακόμη μια φορά επέμενε για τη σημασία προώθησης, ε, μάλλον προόδου σε αυτή την ατυχή υπόθεση. Ε, μόλις χθε μάλιστα παρουσιάσαμε μια νέα πρόταση που περιλαμβάνει δύο νομικές βάσεις. Ε, να πω δύο λόγια και για την Παλαιστίνη όπου έχουμε το θέμα της ενίσχυσης της χρηματοδότησής της για το 2012 μέσω ενός front-loading όπως το λέμε Τώρα δηλαδή εξετάζεται ο προπολογισμό και μέσα στο πλαίσιο τη εκτέλεση του 2011 θα μπορούσε να σα προταθεί και έτσι να ρυθμιστεί ένα τμήμα των προβλημάτων που έχουμε εντοπίσει για αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά τα αποθεματικά πρόεδρε, ε, σημειώνουμε πως ως ήθιστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να στείλει κάποια μηνύματα, αλλά θα ήθελα επίσης ως ήθιστε να θυμίσω ορισμένα σημεία και την σημασία του να μεριμνήσουμε ώστε αυτά τα αποθέματα να μην είναι σε αντίθεση με τις νομικές και πολιτικές δεσμεύσεις και να σέβονται τους, ε, τις γραμμές του προπολογισμού τις οποίες αναφέρονται. Να πω ότι το επίπεδο των πιστώσεων που έχει τεθεί σε αποθυματικό δεν πρέπει να είναι υπερβολικό για να μην εμποδίσει την εκτέλεση του προπολογισμού το πρώτο εξάμεινο του 2012. Να σας πω βέβαια ότι ανησυχούμε ιδιαίτερος λόγω των αποθυματικών για τις διοικητικές δαπάνες που ανέρχονται στα 15,8 εκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχούν στο, σε 317 θέσεις και που μάλιστα στοχεύουν ορισμένες υπηρεσίες της Επιτροπής. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ήδη είχαμε εξετάσει τον περασμένο χρόνο. Ήθελα να επανέλθω εδώ ότι αν θέλετε να διατηρήσετε αυτά τα αποθέματα θα έπρεπε να ομαδοποιηθούν στο επίπεδο της γενικής γραμμής των αμοιβών, των μισθών, για τον απλό λόγο ότι εμείς καθώς είμαστε ένας και μοναδικός ε, εργοδότης δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσει ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες. Αυτό ήθελα λοιπόν να το τονίσω άλλη μια φορά. Και εδώ η διαχείριση θα γινόταν πιο δαπανηρή, αλλά επαναρχόμαστε στα αυτά στην επιστολή σχετικά με την εκτέλεση τη δυνατότητα εκτέλεση και θα τα συζητήσουμε βέβαια και στην Επιτροπή Συνδιαλλαγή. Να επανέλθω επίση ε, για δύο ε, σημεία. Καταρχήν, πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικέ δράσει και δεύτερον, ε, πιστώσει διοικητικέ για τις πιλωτικές δράσεις και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Έχουμε προβλέψει την εφαρμογή μιας, ενός προσωρινού καταλόγου αυτών των ε, προγραμμάτων, αυτών των σχεδίων και ελπίζουμε πως η ανάλυση την οποία κάναμε θα σας φάνηκε χρήσιμη. Επιβεβαιώνουμε την επιθυμία μας για συνεργασία για να φτάσουμε σε μια αποτελεσματική εφαρμογή των πιλωτικών αυτών δράσεων. Και τέλος, όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγχύτρια που φρόντισε ώστε οι διοικητικές δαπάνες που αφορούν το σύνολο των θεσμικών σωμάτων να αποκατασταθεί ή ε, διοικητικέ δαπάνες που σχετίζονται με την προσχώρηση της Κροατίας, διαστατική επιστολή 2012 δεν λαμβάνεται ακόμα υπόψη για αυτή την ανάγνωση της ε, Κομπού, αλλά θα το εξετάσουμε στη διάρκεια της συνδιαλλαγής από ό,τι κατάλαβα. Να πω επίσης πως... Ε, Έχουν μπει στον προπολογισμό οι διαρκητικέ γραμμέ για τα προγράμματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη λειτουργία και ελπίζω πω η, η Γενική Συγγήτρια θα υποστηρίξει αυτό το διάβημα των ειδικευμένων επιτροπών, αν και διαπιστώνω ότι για την κατηγορία 4 δεν υπάρχει πλήρης αποκατάσταση αυτών των γραμμών, πράγμα το οποίο μας δημιουργεί κάποιες ανησυχίες. Στόχος όσον αφορά τους στόχους και τις προθέσεις της Κομπού για αυτό το θέμα. Αυτά ήθελα να πω σύντομα αρχικά. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά θέματα για την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακριβή σας και σύντομη περιγραφή. Μου δίνετε μια πληροφορία που είναι εξωτερικά ενδιαφέρουσα όσον αφορά το ρυθμό κατανάλωσης των πιστώσεων πληρωμών για φέτος, γιατί είδαμε Μάλλον ακούσαμε διάφορα αντιφατικά σχόλια και φήμες. Μάλιστα πριν από κάποιες μέρες η Προεδρία του Συμβουλίου μας έδωσε την ιδέα πως, το, πως οι γραμμές κατανάλωσης ήταν ε, περιορισμένες μετά από τις έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες της αρχής του έτους. Είχαμε επανέλθει σε έναν μέτριο ρυθμό που επιβεβαίωνε την απόφαση που είχε ληφθεί για τον προϋπολογισμό του 2011 ώστε να περιορίσουμε στο 2,91% την αύξηση των ε, πιστώσεων πληρωμών και επιβεβαίωνε και την ψήφο του Συμβουλίου για το 2012 για τις πιστώσεις πληρωμών. Δυστυχώς αυτό που μας λέτε πραγματική εξέλιξη δεν είναι αυτή. Και ότι αντίθετα στα τέλη του έτους κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια συνήθιστη κατάσταση όπου στο τελευταίο διευθυντικό προπολογισμό δεν θα υπάρχουν πλεονάσματα για επιστροφή στα κρατημέλη αλλά επιπλέον πιστώσεις πληρωμών που θα πρέπει να κινητοποιηθούν δεδομένων των αναγκών. Και αυτή η πληροφορία είναι πολύ σημαντική φυσικά για την ψηφοφορία που θα γίνει. Μιλήσατε για το θέμα της βοήθειας στην Παλαιστίνη και το, το συζητήσαμε και στους συντονιστές. Το θέμα είναι υπό εξέλιξη καθημερινή. Πριν από δύο μέρες ενημερωθήκαμε για την απόφαση που έλαβε το Κογκρέσο για να διακόψει την Αμερικανική βοήθεια. 200 εκατομμύρια δολάρια. Εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμού δεν θα εκφραστούμε όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και το περιεχόμενό της, Ένωση. Η Επιτροπή Εξωτερικών θα ασχοληθεί. Αλλά να θυμίσω, το, το θυμίζω μάλλον αυτό που έγινε, ούτως ώστε στην ψηφοφορία που θα γίνει να το έχουμε υπόψη μας. να είναι σαφές ότι η δική μας βοήθεια δεν θέλει να υποκαταστήσει την έλλειψη βοήθειας από άλλους. Εν πάση περιπτώσει θα τεθεί αυτό το θέμα. Πάντως δεν είναι θέμα της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Δεδομένης της σημασίας λοιπόν αυτού του θέματος που είναι υπό εξέλιξη καθημερινά θα πρέπει να το προσέξουμε. και ότι μέσω της κυρίας Άστον αυτή τη στιγμή το, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βαραίνει με όλους τους το κύρος στο πλαίσιο του κουαρτέτου και τα λοιπά και φυσικά αυτό προϋποθέτει και ε, οικονομική συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά τις ανησυχίες για την, ε, τα αποθεματικά, το λαμβάνουμε υπόψη και πιστεύω πως θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση. Κυρία Εισηγήτρια. Κυρία Εισηγήτρια, μπορείτε να μας πείτε τώρα ποια είναι η κατάσταση προετοιμασίας εντός της Επιτροπής του Προπολογισμού για να προετοιμαστεί η ψηφοφορία και βεβαίως να απαντήσετε στα όσα μας είπε και ο Γενικός Διευθυντής. Grazie Presidente, ringrazio anche il Direttore Generale. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Γενικό ο Διευθυντή. Είχαμε μια μακρά συνεδρίαση με τους συντενιστές που ήταν εξαιρετικά χρήσιμη γιατί έτσι ε, μπορέσαμε να τελειοποιήσουμε αυτή την εργασία ε, τη συμβιβαστική συνεργασία που ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Θα έλεγα ότι πάνω κάτω βρίσκουμε μια συμφωνία με την έντονη βούληση να φτιάξουμε μια κοινή θέση του Συμβουλίου σε συνοχή με τα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα, με τα όσα έχουμε ψηφίσει για τα κεντρικά ζητήματα, διατηρώντας κυρίως αυτή την στρατηγική ε, επιλογή, δηλαδή να εστιάσουμε την προσπάθειά μας και τους πόρους μας σε λίγες συγκεκριμένες προτεραιότητες που είναι αυτές τις οποίες υποδεικνύουμε και ως πρώτες προτεραιότητες της στρατηγικής 2020. Ε, ε, συγκεκριμένα και εμείς καταφέραμε να φτάσουμε στη συμφωνία ε, για τα, εκείνα όπου, τα σημεία όπου υπήρχαν αρνητικά περιθώρια και λόγω της, και, την, της στρατηγική σημασία που έχουν, τον, την 1α και την 4, αυτές τις κατηγορίες. Και έπειτα Θέλουμε να εκφράσουμε και τη βούληση να, εκφράσουμε, να χρηματοδοτήσουμε τις προτεραιότητες ε, όπως τις διατύπωσαν οι ομάδες και οι ειδικευμένε επιτροπές. Και για αυτές στο Κοινοβούλιο θα υπάρξει αίτημα να ξεπεράσουμε και την πρόταση την οποία επεξεργάστηκε η Κομισιόν τον περασμένο Απρίλιο και να ζητήσουμε τη χρήση της ευελιξίας 30 ε, εκατομμυρίων σε αυτό το τίτλο. Προτεραιότητες είναι το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, η ΚΑΠΑ στις δύο γραμμές και το το lifelong learning, για το οποίο θα ζητήσουμε σημαντική αύξηση πέρα από την πρόταση της Κομισιόν για την Κατηγορία 4, η προσπάθεια είναι ακόμη πιο μεγάλη, γιατί η αρχική αρνητική εικόνα ήταν ήδη πολύ σημαντική. 153 εκατομμύρια στην πρόταση της Επιτροπής. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια αξιοσημείωτη για να καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε τις προτεραιότητες ε, των χωρών της Μεσογείου, το είχαμε ήδη αυτό συμπεριλάβει και στην εντολή για τον τριμερή διάλογο και παρουσιάζουμε και μια συμφωνία με 100 εκατομμύρια παραπάνω για την Παλαιστίνη. Και αυτό ήταν ένα σημείο το οποίο είχαμε ε, χρησιμοποιήσει στην εντολή για τον τριμερή διάλογο. Εφόσον υπάρξει λοιπόν Καταλήξαμε δηλαδή στα 208 εκατομμύρια ευελιξία για αυτές τις δύο κατηγορίες. Βλέπουμε λοιπόν πως πρόκειται για μία συνεπή γραμμή με βάση τις προτεραιότητες που είχαμε ήδη επιλέξει και συνεπή με το πνεύμα της ε, προσπάθειας για, σύσταση, για σύνταξη ενός προπολογισμού πιο συνεπούς και πιο ισχυρού τη στιγμή των διαπραγματεύσεων. Και έτσι καταφέραμε να εκφράσουμε ξεκάθαρα τις προτεραιότητες και τις βούληση όχι μόνο της Επιτροπής Προπολογισμών αλλά και όλων των επιδικευμένων επιτροπών και των πολιτικών ομάδων που συμμετείχαν εξ αρχής στην διαβούλευση να εκφράσουμε δηλαδή την πραγματική βούληση του Κοινοβουλίου στις πολιτικές που θέλει να χρηματοδοτήσει το 2012. Το μέσο των πιλωτικών προγραμμάτων και των προσκευαστικών δράσεων ε, ε, χρησιμοποιήθηκε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πάντοτε για χρηματοδότηση ευαίσθητων προτεραιοτήτων μέσα στη στρατηγική 2020 και για να υπάρξει και μια αντιστάθμιση κατά κάποιο τρόπο, γιατί ξέρουμε πως δεν υπήρχαν πάντοτε οι απαραίτητοι πόρες στο εσωτερικό των διαφόρων κατηγοριών και ήταν πολύ χρήσιμη η δουλειά που κάναμε με την Επιτροπή, ότι δηλαδή είχαμε ένα feedback ε, για το κατά πόσο όλα αυτά προτείναμε ήταν εφικτά από τεχνικής άποψης. Εισάγαμε και αυτό ήταν ε, βασική βούληση όσον αφορά την ε, νομική βάση για το τις προτεραιότητές μας και θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι την πρότασή του να μπουν τα αποθυματικά σε μια γενική γραμμή και όχι υπό τις μεμονωμένες γενικές διευθύνσεις. Θα ήθελα να τον καθησυχάσω λοιπόν υπό την έννοια ότι συμφωνώ με την πρότασή του. Επίσης είμαι πολύ ικανοποιημένη με τα όσα μας είπε ο Διευθυντής για το επίπεδο των πληρωμών, ότι είναι κάτι για το οποίο συζητήσαμε πολύ κυρίως στο ιστορικό των ε, συντονιστών, γιατί είναι κάτι επί το οποίο διχαστήκαμε και ως ομάδες. Ανέκαθεν λέγαμε ότι οι πληρωμές και οι υποχρεώσεις θα έπρεπε να εφαρμόζονται περισσότερο με τη στρατηγική, υπάρχει στρατηγική για τις υποχρεώσεις, αλλά για τις πληρωμές διχαστήκαμε γιατί Είχαμε αντιφατικές πληροφορίες όσον αφορά την πραγματική ανάγκη καταβολής αυτών των πληρωμών. Τέλος όμως και εξ αρχής το προτείναμε να προχωρήσουμε με συνοχή σε αυτή την εντολή στον τρίλογο, δηλαδή να θεωρήσουμε ως μίνιμουμ, ως το τελικό όριο το επίπεδο των πληρωμών που προτείνει η Κομισιόν και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω θα φτάσει ε, η συμφωνία με μεγάλη πλειοψηφία και να πω ότι είμαι ικανοποιημένη που βλέπω ότι αφού έγινε μεγάλη προσπάθεια για να γίνει μια καλή πολιτική επιλογή για τον προτεραιοτήτων μας, προσπαθήσαμε επίσης να συμφωνήσουμε για μια σοβαρή ε, στρατηγική γραμμή, ώστε να μας, ε, να μην υπάρξει μεγάλος χώρος για τις διαπραγματεύσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε κοντά στο τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε, στις δικές μας προτεραιότητες. Και είμαι ικανοποιημένη για το γεγονός ότι εξ αρχής παρουσιάσαμε μια γραμμή εμπιστοσύνης με, στην ε, Κομισιόν. Και αυτό ήταν μια καλή ένα, ένα καλό σημείο κίνηση για τις διαπραγματεύσει που θα αρχίσουν στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο Χωσέ Μανουέλ Φερναντές, μπορείτε να μας ε, κάνετε τη δική σας παρουσίαση. Να μας παρουσιάσετε δηλαδή τις ε, προτάσεις σας για την ψηφοφορία. Ε, Τάχει το προπολογισμό του Κοινοβουλίου, αλλά επίσης να πείτε κάποια λόγια για τους προπολογισμούς των άλλων θεσμικών οργάδων. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ να ξεκινήσω από τα άλλα θεσμικά όργανα. Ο στόχος είναι τα θεσμικά όργανα να έχουν το μήνυμα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, να καλύψουν τις αρμοδιότητές τους, να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και τις νέες αρμοδιότητες που τους αναθέτει η συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό και κάναμε μια δουλειά συγκεκριμένη όσον αφορά ε, τα θεσμικά όργανα και έτσι να υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι τόσο στο Κοινοβούλιο για τις επιπλέον ε, προσπάθειες που πρέπει να κάνει και γι' αυτό κάνουμε και μια μερική αποκατάσταση εν γέννη στο σύνολο των ε, θεσμών με την εξαίρεση του ΔΕΚ. κάνουμε γενική αποκατάσταση της πρότασης και για το ΔΕΚ κάνουμε πλήρη αποκατάσταση που γιατί είναι μικρό όργανο. Σε σχέση με το Κοινοβούλιο, αυτό ε, περάσαμε χωρίς την Κροατία και χωρίς τους 18 νέους ε, βουλευτές έχουμε περάσει σε 1,9 αύξηση με την Κροατία και τους νέους ε, βουλευτές. 70 εκατομμύρια έχουμε περικόψει. Εάν συγκρίνουμε την αύξηση και την ενημέρωση του προπολογισμού του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου είναι 0,8%. Χωρίς την Κροατία και τα νέα μέλη, αυτός είναι, αυτή είναι η αύξηση. Και θα πρέπει να κάνουμε σύγκριση μεταξύ συγκρίσιμων μεγεθών. Είμαστε στη γραμμή κάτω από το στόχο που έχει χαράξει ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι και η επιστολή που μας έστειλε σε όλους τους θεσμούς, σε όλα τα θεσμικά όργανα. Και όσον αφορά το Κοινοβούλιο και το... τις τροπολογίες που ολοκληρώνουμε, δύο προγράμματα τα αφήσαμε. Όσον αφορά τα κονδύλια, το πιο σημαντικό ήταν εκείνο το πρόγραμμα που σχετιζόταν με ένα πιλωτικό πρόγραμμα που πρότεινε η ΑΦΕΤ. Ένα πρόγραμμα λοιπόν το οποίο εγκαταλείψαμε. Τώρα, σε σχέση με τον οίκο της ιστορίας που ήδη έχει ένα αποθεματικό και την παρουσίαση του σχεδίου που είχαμε ήδη εγκρίνει την άνοιξη υπάρχει μια καινοτομία που για μας είναι σημαντική και που έρχεται να ικανοποιήσει το σύνολο των ομάδων και έχει να κάνει με την ανάκτηση από πλευράς ε, θεσμικής ε, των στόχων αυτού και μάλιστα ε, είμαστε ικανοποιημένοι με την επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής που υποστηρίζει το σχέδιό μας. Σε σχέση με την παρουσίαση των τροπολογιών, μάλλον σε σχέση με τα θέματα εκείνες τις τροπολογίες που μπορεί να γίνουν ή όχι δεκτές. Εν γέννη, πρόκειται για τροπολογίες που έχουν να κάνουν με το καταστατικό του Ευρωβουλευτή. Δεν θα ξαναψηφιστούν και εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία για να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες, τις πολιτικές και τους Κεώδης για την ε, προσπάθεια που έκαναν. Να ευχαριστήσω και το Προεδρείο γιατί φτάσαμε σε μια συμφωνία εξαιρετική που θα υποχρεώσει ε, να γίνουν ε, διαπιστωτικές αλλαγές στο Κοινοβούλιο. Στην πράξη με τους νέους κανόνες που θα ισχύσουν για την διερμηνία καταφέραμε να κάνουμε μια επιπλέον εξοικονόμηση 10 εκατομμυρίων ευρώ με τη μετάφραση 11 εκατομμύρια εξοικονόμηση γιατί σταματά να είναι αυτόματη η μετάφραση σε όλες τις γλώσσες και να είναι ξεκάθαρο αυτό η αρχή είναι η αρχή της πολυγλωσσίας αυτή δεν αμφισβητείται ποτέ δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί γιατί εξάλλου εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση γιατί κατόπιν αιτήματος μπορούν να γίνονται οι μεταφράσεις. Θα έλεγα ότι το Ευρωκοινοβούλιο προχωρά σε μια νέα φάση σύμφωνα με τις αρχές της στρατηγικής 2020. Θέλουμε δηλαδή βιωσιμότητα και ενοτομία που να οδηγεί σε εξοικονόμηση και όλα αυτά να γίνουν με ευφυή τρόπο. Οι προτεραιότητες της στρατηγικής 2020, ευφυής ανάπτυξη για όλους και βιώσιμη ανάπτυξη είναι εδώ σαφή. Και γιατί πολλές από τις νέες ε, αρμοδιότητες ε, οδηγούν στο να μπουν νέοι πάλι στις, ε, στα θεσμικά όργανα και εδώ αποδεικνύεται ότι με λιγότερους πόρους μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δράσεις. και να καλύπτουμε περισσότερες αρμοδιότητες. Αποτελεσματικότερη δηλαδή και αποδοτικότερη η χρήση των διοικητικών μας δομών. Εξάλλου αυτό περιμένουν από εμά και οι πολίτες, να απαντήσουμε με ποιότητα. Νομοθετική αριστεία είναι ένας στόχος ο οποίος ε, εξακολουθεί επίσης να ισχύει και παρουσιάζουμε έναν, υποβάλλουμε μάλλον όλα τα θεσμικά όργανα, υποβάλλουν προϋπολογισμούς που στην ουσία ε, ε, αντιστοιχούν σε αρνητική ανάπτυξη γιατί είναι πολύ κάτω από τον πληθωρισμό. Οι βουλευτές επίσης συμβάλλουν ώστε αυτό να γίνει δυνατό, όπως και οι υπάλληλοι του θεσμικού οργάνου είναι ένας τρόπος ώστε να είμαστε στην ίδια γραμμή ε, με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες σε αυτή τη τόσο δύσκολη φάση που διανύει ολόκληρη η Ευρώπη και που ευχόμαστε να είναι περαστική. Σας ευχαριστούμε και θα ήθελα απλώς να επιμείνω σε ένα σημείο. Υπάρχει κάποιος που θέλει να πάρει το λόγο. Ο συνάδελφος ε, κύριος Βόγκαν. Παρακαλώ. Λοιπόν, πρόεδρε, απλά να απαντήσω σύντομη, συντομία ε, στη τελευταία ερώτηση του κύριου Φερνάντες. Όπως είπε και πολύ ορθά, Υπάρχει συμφωνία ευρεία πλέον για τα πιο πολλά ζητήματα για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου και για τους άλλους ε, θεσμικούς οργανισμούς. Συμφωνούμε, για παράδειγμα, ότι θα πρέπει εν μέρη να επαναφέρουμε τον προπολογισμό τους, ή άλλως θα έχουν πρόβλημα στη λειτουργία του στο μέλλον. Για τα άλλα θέματα που αναφέρθηκαν τώρα, νομίζω ότι ξέρουμε ότι λάβαμε διάφορες εγγυήσει για τον οίκο της ιστορίας και σε ό,τι αφορά την ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου Πρόσφατα λάβαμε τέτοια στοιχεία, καλό θα είναι να τα διαβάσουμε. Νομίζω ότι πολλοί συνάδελφοι έλαβαν πολλέ πληροφορίες. Τώρα, σε τι αφορά τα άλλα ζητήματα για τα έξοδα ταξιδίου, έχουμε μείωση 5% και υπάρχει συμφωνία τώρα για το πάγωμα των μισθών των επιδομάτων. Νομίζω ότι υπάρχει γενική συμφωνία να παγώσουν τα GEA για το επόμενο έτος. Οι σοσιαλιστές θα ήθελα να πάνε λίγο παραπάνω και να, και να παγώσουν όλα τα, όλα αυτά τα ποσά για το επόμενο έτος. Εμείς θα εξετάσουμε τον δεχόμενο να καταθέσουμε σχετικές ε, τροπολογίες. Μπορεί να μην τις κρίνετε παραδεκτές γιατί το, οι σοσιαλιστές λένε να μην παγώσουν μόνο τα GA, αλλά και Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι. Αναφέραμε ε, διαμακρών το πρόβλημα αυτό συνάντηση των συντονιστών και θα ήθελα να πω το εξή. Όσο αφορά τις ενδεχόμενε τροπολογίες, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, από όσο γνωρίζω, τυχόν ε, τροπολογίες που θα αφορούν τις αποδοχές των βουλευτών, των υπαλλήλων μάλλον. Δεν έχουμε την ε, νομική αρμοδιότητα. Αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό και επικυρώθηκε από την απόφαση του δικαστηρίου που καταδικάζει την απόφαση του Συμβουλίου που είχε, ε, δεν είχε εφαρμόσει το καταστατικό και είχε παγώσει τα επιδόμετα. Για όλες τις άλλες διατάξεις που συνδέονται με το καταστατικό, αλλά δεν αφορούν τις αποδοχές, δηλαδή τις αποζημιώσεις και άλλες. Και αυτή είναι η άποψη της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου η απόφαση να πόκειται στο Προεδρείο. Αλλά βεβαίω η Ολομέλεια μπορεί να το ακυρώσει. Δηλαδή το Προεδρείο δεν είναι, στο, το Προεδρείο δεν έχει την ε, κυριαρχία. Την κυριαρχία την έχει η Ολομέλεια. Και για να μπορέσει να αποφανθεί η Ολομέλεια στη δική μας διαδικασία για τον προπολογισμό θα πρέπει οι τροπολογίες να ε, υποβληθούν στη δική μας επιτροπή. Εάν υπάρχουν ε, τροπολογίες για αυτή την κατηγορία είναι τροπολογίες που αποκλίνουν από την πολιτική συμφωνία γιατί υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ Κοκομπού και Προεδρία. Εάν λοιπόν αυτές οι τροπολογίες θα ε, υποβληθούν στην ψηφοφορία και στη συνέχεια μπορούν να πάνε στην Ολομέλεια. Και θα είναι το Κοινοβούλιο, το σώμα το οποίο θα αποφασίσει για την νομική του εγκυρότητα στην Ολομέλεια. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πολιτικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Και θα ήθελα να προσθέσω και μια τελευταία παρατήρηση και συγκεκριμένα προς ενημέρωση του αδελφού Ράιμερ Μπέγκε, ο οποίο είχε προσκληθεί στη συνεδρίαση των συντονιστών, αλλά μπορούσε να συμμετάσχει και καλύτερα πράγματα να κάνει. Η Φραντσέσκα Μπαλζάνη είπε ότι προσανατολισόμαστε προς μια πολιτική συμφωνία η οποία θα καταλήξει στην υπέρβαση του πλαφών για τις κατηγορίες 1α και 4 για σχετικά μικρά ποσά. Και η πολιτική ιδέα έγκυται στο, ε, το οποίο κάναμε και την περασμένη χρονιά, δηλαδή να μην ψηφίσουμε τις ορπολογίες με αστερίσκο, διατυπώς, ενα τρόπο στον οποίο είχαμε προσφύγει και πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας και από νομική άποψη ήταν κάπως αμφίβολος πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας και είναι ακόμη περισσότερο μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και να ανταυτού να προτείνουμε στις τροπολογίες μας σύμφωνα με αυτό που έκανε για πρώτη φορά σχέδιο προπολογισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μία από τις κατηγορίες να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα πλεονάσματα κινητοποιώντας το εργαλείο ευελιξίας, το μέσο ευελιξίας. Άρα είναι ο συγκητής για την διοργανική συμφωνία, ο οποίος θα πρέπει να χρωματοδοτήσει για τη διαδικασία για να δούμε πώς μπορούμε, εφόσον συμφωνεί βεβαίως, σε εύλογο χρόνο, να ψηφίσουμε την έκθεσή του ταυτόχρονα με τον προπολογισμό, όπως ε, το κάναμε θα το κάναμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Πακοσμιοποίηση και όπου έχουμε ταυτόχρονα ανάγκη μιας ε, ψηφοφορίας ε, για τον προπολογισμό υπό τη στενή έννοια και μιας ε, ψηφοφορίας για την έκθεση του Ράιμερ σύμφωνα με την, σε σχέση με τη διοργανική συμφωνία και σύμφωνα με την Οργανική Συμφωνία. Ε, ίσως ε, στη μεσημεριανή παύση μπορούμε να διευκρινίσουμε περισσότερο αυτή τη διαδικασία για να εξασφαλιστούμε ότι όλοι αποδέχονται αυτή την οδό. Αγαπητοί συνάδελφοι, εάν δεν θέλει κανεί άλλο να πάρει το λόγο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γενικό Διευθυντή Λύεται συνεδρίαση και θα σας δίνω ραντεβού στις 3 το απόγευμα με τις κάρτες σας της ψηφοφορίας, φυσικά, γιατί βεβαίως θα τις χρειαστούμε και φυσικά όλους τους πίνακες της ψηφοφορίας και όλα τα έγγραφα. Λύεται συνεδρίαση. Ευχαριστώ.